του Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015 και έχει το λόγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Τούσκ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου αντιμετώπισε όλες τις σημαντικές κρίσεις που γνώρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015. Είτε μιλάμε για την προσφυγική κρίση και τους μετανάστες, είτε μιλάμε για την μεταρρύθμιση της ΟΝΕ. Σε όλες αυτές τις συζητήσεις σημειώσαμε πρόοδο, αλλά σίγουρα όχι αρκετή πρόοδο. Αναμφίβολα λοιπόν το 2016 θα επισκιαστεί από τις προκλήσεις αυτές. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται από τις κρίσεις αυτές. Και αυτή τη στιγμή δοκιμαζόμαστε σε όλα τα πιθανά μέτωπα ταυτοχρόνως. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να πω ξεκάθαρα και με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να σταματήσω να εργάζομαι μέχρι να βρούμε λύσεις για όλες αυτές τις προκλήσεις. Η δύναμή μας αντλείται από το ότι είμαστε ενωμένοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να παραμείνουμε ενωμένοι και αυτό ήταν ο βασικός μου στόχος και το 2016. Αξιότιμα μέλη, Α ξεκινήσω με το ζήτημα της μετανάστευσης και με το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης και με την υπαρξιακή αυτή κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. όπω τα θυμάστε, για πάρα πολλού μήνε, ήδη δηλαδή από την αρχή τη προσφυγική κρίση τόνισα ότι ε, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική από την προστασία των συνόρων. Αυτή είναι μια προϋπόθεση εκ των ΟΚΑΝΕΦ προκειμένου να έχουμε οποιαδήποτε στη συνέχεια με την εστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν καταφέρουμε να επιτηρήσουμε παρκώς τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ως πολιτική κοινότητα θα αποτύχουμε. Μετά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μπορούμε να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Οι συζητήσεις των αρχηγών κρατών κυβερνήσεων επικεντρώθηκαν στους τρόπους και στα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε την προστασία των εξωτερικών συνόρων και όλοι οι ηγέτες αναγνώρισαν ότι η προστασία του Σέγγεν περνά από δύσκολες αποφάσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό συμφωνήσαμε να εξετάσουμε πολύ γρήγορα την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένη τη νέα ιδέα για μια Ευρωπαϊκή Συνοριακή συνοριοφυλακή και αυτοφυλακή. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Ολλανδικής Προεδρίας και θα έχουμε μέχρι τον Ιούνιο κάποια συμφωνία. Το γεγονός ότι έγινε δεκτό από την Ελλάδα να χρησιμοποιηθεί η νέα δύναμη ταχείας επέμβασης της Frontex αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολονότι έχουμε πρόοδο στο πολιτικό επίπεδο, στην πράξη υπολοιπόμεθα ακόμα πολύ. Όσον αφορά τα hot spots, όσον αφορά την εξέταση ασφαλείας των τρίτων χωρών και όσον αφορά επίσης το ζήτημα της μετεγκατάστασης και των επιστροφών. Επίσης έχουμε ένα σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την Τουρκία, το οποίο ακόμα όμως δεν έχει αποδώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Συμφωνώ επίσης μετά όσο είπε ο Πρωθυπουργός Ρούτε, ότι έχουμε μόνο δύο μήνες διαθεσή μας προκειμένου τα πράγματα να αρχίσουν να λειτουργούν. Τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε για την περίοδο των Χριστουγέννων δεν είναι θαρρυντικά. Πάνω από 2.000 αφήξεις είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ημερήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Frontex. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα είναι τελευταία ευκαιρία για να δούμε τελικά αν η στρατηγική μα λειτουργεί στην πράξη. Και αν δεν λειτουργεί η στρατηγική αυτή, τότε θα αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικέ συνέπειε, όπω η κατάρρευση του Σέγγεν. Σίγουρα λοιπόν δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία τέτοια εναλλεκτική στη στρατηγική μας. Γι' αυτό το λόγο καλό τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την ε, στρατηγική που έχουμε για το μεταναστευτικό ζήτημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε τώρα στο ζήτημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Δεκέμβριο οι ηγέτε ε, κρατών και κυβερνήσεων κάνανε μια πλήρη συζήτηση όσον αφορά το ζήτημα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Πρωθυπουργό Κάμερον εξέθεσε λεπτομερώ ε, τη θέση του, ιδίω όσον αφορά τα επιδόματα και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Είπε ότι ε, θέλει να προβλέπεται μια περίοδο τεσσάρων ετών παρανομή στο Ηνωμένο Βασίλειο και είπε ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτό οι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεντρωθήκαμε επίσης σε συγκεκριμένα ζητήματα και είπαμε επίσης ότι θέλουμε να βρούμε και κάποιες συμβαστικές λύσεις. Βασιζόμενοι λοιπόν στην πρώτη αυτή θετική συζήτηση που κάναμε, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε εκ νέου προκειμένου να βρούμε λύσεις και για τα τέσσερα αυτά ζητήματα τα οποία έθιξε ο Πρωθυπουργό Κάμερον οι σχέσει με τι χώρε τη Ευρωζώνη, το ζήτημα τη κυριαρχία, το ζήτημα τη ανταγωνιστικότητα, το ζήτημα τη ελεύθερη κυκλοφορία, καθώ επίση και των κοινωνικών παροχών. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο και αυτό ήδη έχει γίνει και για τα τέσσερα αυτά ζητήματα και εργάζεται επίση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ζητήματα αυτά. Μέχρι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου θα έχω αποβάλει και εγώ συγκεκριμένε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ το Ηνωμένο Βασίλειο, προτάσει που θα πάνε προ όλου του αρχηγού κρατών κυβερνήσεων. Για άλλη μια φορά θέλω να πω ότι από την αρχή των διαπραγματεύσεων αυτών ήμουν απόλυτα σαφή. Δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα συμβιβασμό σε θεμελιώδη δικαιώματα όπω η ελεύθερη κυκλοφορία και η ε, μη διακριτική μεταχείριση. Παράλληλα, θα κάνω κάθε τι το δυνατό προκειμένου να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση και για την Βρετανική πλευρά από σήμερα τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ουσιαστικά δεν μπορούν να προβλεπτούν. Είναι όλο και περισσότερο απρόβλεπτα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα και γι' αυτό το λόγο θα εργαστώ πολύ αποτελεσματικά για να έχουμε ήδη το Φεβρουάριο μια συμφωνία. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, αλλά πιστεύω ότι είναι ακόμα δυνατό να πετύχουμε μια τέτοια λύση. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το ζήτημα της καταπολέμησης τρομοκρατίας υπό το φως τρομοκρατικών επιθέσεων του Παρισίου. Οι τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις ενίσχυσαν τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσει τρομοκρατία. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν ότι θα πρέπει να υπάρχει πλέον μια συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τους ξένους μαχητές μέσω του Σέγγεν και μέσω της Ευρωπόλ, αλλά και μια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών. Επίσης, ε, θα πρέπει να γίνονται κοινέ αναλύσεις όσον αφορά το ζήτημα της ε, της ασφάλειας για να καταφέρουμε να αποφύγουμε μελλοντικέ τέτοιε επιθέσεις. Ήδη η Ευρωπόλ μας λέει ότι υπάρχει μια ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τους ξένους μαχητέ, ιδίως μέσω του νέου κέντρου αντιτρομοκρατία τη Ευρωπόλ, όπου κάθε κράτος μέλος πλέον συνεισφέρει με, επιπλέον δεδομένα. Χωρί συνεργασία αυτή δεν θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την απειλή. Και Ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετέ πιθανότητε και για νέε τρομοκρατικέ επιθέσει. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ζητώ από όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν πλήρω. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης αποτέλεσε ευκαιρία για τους ηγέτες να αξιολογήσουν το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την Ενεργειακή Ένωση και τη δημιουργία μάλλον της Ενεργειακής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τη διασύνδεση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και των αγορών φυσικού αερίου, εμπλέκοντας περισσότερο κράτη-μέλη τα οποία ήταν περισσότερο απομονωμένα μέχρι σήμερα. Ω ε, Πολωνό Πρωθυπουργό προσπάθησα να προωθήσω ιδιαίτερα την ιδέα τη Ενεργειακή Ένωση και χαίρομαι πάρα πολύ τώρα και με το νέο μου αξίωμα που έχει επιτευχθεί πρόοδος, αλλά περισσότερα πράγματα πρέπει να γίνουν ακόμα. Ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προωθηθεί όλη η απαιτούμενη νομοθεσία, ιδίω όσον αφορά και το ζήτημα της διαφάνειας για τι αγορές φυσικού αερίου. Όσον αφορά την Ενεργειακή Ένωση, οι αρχικοί κρατών κυβερνήσεων κάνανε μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το σχέδιο Nord Stream 2. Ορισμένοι επέκριναν τον το νέο αυτό σχέδιο και επίσης συζητήσαμε τις προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν ε, στα πλαίσια μεγάλων έργων ενεργειακών υποδομών. Είπαμε ότι οποιαδήποτε τέτοια νέα ενεργειακή υποδομή θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. Και είπαμε επίση ότι υπάρχει και μια προφανή υποχρέωση όλα τα ενεργειακά αυτά έργα να συνάδουν με τη συνολική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένη στις τρίτη δέση μέτρων για την ενέργεια. Αυτέ είναι ξεκάθαρε προποθέσει προκειμένου να υπάρχει υποστήριξη από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από, από οποιοδήποτε κράτο μέλο. Πολιτική ή οικονομική υποστήριξη. Εναπόκειται τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει περισσότερο τα απαιτούμενα αυτά νομοθετήματα. Το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν ξεκάθαρο και ουσιαστικά κινείται στην κατεύθυνση που κινείται και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Επίσης, οι ηγέτες συνεχάρισαν τον πρόεδρο Ολόν, τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας για τη διοργάνωση της COP21 και το γεγονός ότι καταλήξαμε σε μια παγκόσμια πλέον συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Συμβούλιο να αξιολογήσουν πλήρω τι επιπτώσει τη Συμφωνία των Παρισίων όσον αφορά τη δική μα πολιτική για την ενέργεια και για το ενεργειακό μείγμα. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι και το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντιμετώπισε το ζήτημα των οικονομικών προκλήσεων. Οι ηγέτες είπαν ότι θέλουν να συνεργαστούν περισσότερο προκειμένου να ολοκληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση βασιζόμενη στην έκθεση των πέντε προέδρων. Μολονότι αυτή τη στιγμή ασχολούμεθα πολύ βέβαια με την προσφυγική κρίση, δεν γίνεται να ξεχάσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί και να βελτιωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων είπαν ότι θα πρέπει να σημειθεί η πρόοδο σε πάρα πολλού τομεί, συμπεριλαμβανομένη και τη Τραπεζική Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβαθύνουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, καθώς επίσης και την ψηφιακή αγορά και να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε επίσης και την Ένωση Κέφαλε Αγορών. Αγαπητοί συνάδελφοι, τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλοί οι οποίοι προωθούν μια πολύ απεσιόδοξη προσέγγιση όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ε, Ευρωπαίοι θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά θα πρέπει να έχουμε και εμπιστοσύνη στα πιστεύω μας και στις αξίες μας. Πολύ συχνά μου υπενθυμίζουν ε, μια πολύ σημαντική παρατήρηση που είχε γίνει ότι ο πολιτισμός ουσιαστικά πέθανε λόγω αυτοκτονίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να κάνουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να τροποποιήσουμε την παρούσα κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τούς. Και τώρα το λόγο έχει ο πρόεδρος κύριος Γιούγκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Μετά τις πολύ καλά διαλεγμένες λέξεις του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έπρεπε να συνοψίσω με δύο λόγια τα συμπεράσματα, η μετανάστευση, η τρομοκρατία, η ΟΝΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, θα έλεγα ότι όλα αυτά αντικατοπτρίζουν πλήρως μια Ευρώπη σε πολλαπλές κρίσεις. Πολλής λόγος έγινε τους τελευταίους μήνες για την ελληνική κρίση, για την κρίση των προσφύγων και για άλλες κρίσεις. Στην πραγματικότητα η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια συγκυρία πολλαπλών, περίπλοκων κρίσεων που έρχονται και έξωθεν και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και που σημειώνονται ταυτόχρονα. Σαφέστατα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και καλούμαστε να ξεπεράσουμε την εθνική οπτική γωνία και να ξαναβρούμε το πνεύμα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, την αλληλεγγύη του. Μπορούμε να το κάνουμε εάν το επιθυμούμε μπορούμε να κομίσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση υπεύθυνη και αλληλέγγυα στις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε. διότι περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σημαίνει ότι θα έχει περισσότερες δυνατότητες κάθε χώρα να ξεπεράσει την κρίση που αντιμετωπίζει. Έτσι κάναμε και στο παρελθόν και γι' αυτό είχαμε την ενιαία αγορά και γι' αυτό δημιουργήσαμε τον χώρο Σέγγεν. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να ε, συμπληρώσουμε το πάζλ με τα τελευταία ε, κομμάτια και να τελειοποιήσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επίγουσας προσφυγικής κρίσης. Αν είχαν όλα αυτά υλοποιηθεί, σήμερα θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο όταν ακούω να λένε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην προσφυγική κρίση θέλω να απαντήσω ότι αυτό είναι ψευδές και αληθές ταυτόχρονα. Είναι ψευδές διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με αγαστό τρόπο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κομίσει όλα τα στοιχεία απάντησης που είναι απαραίτητα και είναι αληθές από την άλλη γιατί όλα αυτά θα γίνουν πραγματικότητα όταν τα κράτη-μέλη από τα λόγια περάσουν στις πράξεις. Ορισμένοι πολύ γρήγορα θέλησαν να επικρίνουν την Ένωση της Βρυξέλλες όπως μας λένε και λένε ότι πρέπει η Ένωση και οι Βρυξέλλες να κοιταχθούν στο καθρέφτη. Όμως οι Βρυξέλλες είναι επίσης και εκείνοι και οι ίδιοι. Βρυξέλλες είναι και τα κρατημέλη και οι κυβερνήσεις αυτών. Η έλλειψη δράσης μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη υιοθέτηση δεσμεύσεων εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως το υπογράμμισε το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη πρέπει να ρυθμίσουν τα θέματα της επανεγκατάστασης. Όλα αυτά είναι αποτελεσματικά εργαλεία και θα πρέπει να υιοθετηθούν για την ευρωπαϊκή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Και καλό για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπλέψει μαζί μας για να προχωρήσουμε ε, και να έχουμε Ευρωπαϊκό Σώμα Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Κοινά σύνορα, κοινή διαχείριση. Εάν δεν το συνειδητοποιούμε, η Σέγγεν δεν θα επιβιώσει. Σε μια Ευρώπη με τα παλαιά σύνορα, μια Ευρώπη που δεν γνώρισαν αν είναι σήμερα, σε αυτήν θα επιστρέψουμε δυστυχώς. Ε, ε εγώ θα ήθελα να μην αλλάξει αυτό, δηλαδή οι νέοι που δεν έχουν γνωρίσει την παλιά Ευρώπη με σύνορα να συνεχίσουν να μην την γνωρίζουν. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ε, οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι που διασχίζουν τα σύνορα καθημερινά θα χαίρονταν με την κατάρρευση του χώρου Σέγγεν. Ούτε οι μεταφορικές επιχειρήσεις θα χαίρονταν, γιατί θα σημείωναν πολύ σημαντικές οικονομικές απώλειες με την επανεισαγωγή και επαναθέσπιση των συνόρων. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη γίνονται 26 εκατομμύρια ταξίδια αεροπορικά για επιχειρηματικούς λόγους, πάρα πολλά εκατομμύρια μεταφορών. Όλα αυτά στοιχίζουν. Η τιμή, το τίμημα του να μην έχουμε χώρο Σέγγεν είναι εξαιρετικά υψηλό. Είναι ένα πρόγραμμα κατά της ανάπτυξης και κατά της απασχόλησης το να μην υπάρχει Σέγγεν και πρέπει να κάνουμε το παν για να διασώσουμε το χώρο Σέγγεν γνωρίζοντας ότι όλα αυτά είναι εφικτά μόνο με μια ευρωπαϊκή πολιτική. Και γι' αυτό, λίγαν συντόμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις για την αναθεώρηση των κανονισμών του Δουβλίνου και των κανόνων του Δουβλίνου. Κύριε Πρόεδρε, αν πρόκειται για την ε, φύλαξη των συνόρων, δεν αρκεί να δούμε το θέμα μόνο από τη δική μας πλευρά, αλλά θα πρέπει να δούμε τα σύνορα τα οποία μοιραζόμαστε με τους άλλους, να τα δούμε και από τη δική τους ε, πλευρά. Και χρειαζόμαστε πραγματικά μια πεισματική, προσιλωμένη, καθημερινή εργασία. Δεν χρειαζόμαστε μόνο δηλώσεις πρόθεσης, αλλά πολύ συγκεκριμένη εργασία και διατύπωση κοινών ε, προτύπων. Και το εξίσου επίμονα συνεργαζόμαστε με την ε, Τουρκία η Τουρκία πραγματικά έκανε τα πρώτα θετικά βήμα για ένα κοινό πρόγραμμα δράσης. Ε, για παράδειγμα, θέσπισε μια υποχρέωση θεώρησης εισόδου για τους ε, μετανάστες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, ε, απομένουν πολλά πράγματα να γίνουν προκειμένου να μειωθεί αισθητά η ροή των προσφύγων. Ε, θα πρέπει το κοινό πρόγραμμα δράσης ε, τάχιστα να εφαρμοστεί. Ε, δεν έχω τίποτα εναντίον εκείνων οι οποίοι, εμφανίζουν, οι οποίοι κάνουν κάποιες δηλώσεις οι οποίες παράγουν θετικά αποτελέσματα στο Παρίσι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκε σκληρά για μια συμφωνία η οποία ήταν νομικά δεσμευτική και φιλόδοξη. Ωστόσο η πραγματική εργασία βρίσκεται μπροστά μας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά ώστε να γίνουν νέα βήματα. Εν τω μεταξύ, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι του 2020. Όσον αφορά τη σχέση του Ενωμένου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε μια οικοδομητική ε, συζήτηση με την Βρετανική κυβέρνηση και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπα τότε. Ε, κανένα από τα τέσσερα αυτά θέματα είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουμε και θα το προσεγγίσουμε με μεγάλη σεβαρότητα. Ωστόσο, επιτρέψατε μου να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπα προηγουμένω, θέλει μια έντιμη συμφωνία με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία είναι ισχυρότερη εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρότερη με τη Μεγάλη Βρετανία. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει επίση η συμφωνία να είναι δίκαιη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με του εκπροσώπου του Συμβουλίου στην κατεύθυνση αυτή. Και θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να ολοκληρώσω ε, αποτείοντας ε, τιμή στο έργο αυτού του Κοινοβουλίου γιατί εδώ και 12 μήνες ε, συμμετέχω εδώ και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι παράγονται θετικά επιτελέσματα από αυτό το σώμα. Το Κοινοβούλιο στήριξε την Επιτροπή του ώστε να παράξει θετικά αποτελέσματα. Όταν, χρειάζεται ευελιξία, όταν χρειάστηκε ευελιξία για τις νέες μας προτάσεις και αποτελεσματικότητα, το Κοινοβούλιο στάθηκε στο πλευρό μας και έχω την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει στο πνεύμα αυτό το κοινοβούλιο, τις προσπάθειές του αυτό το έτος και, τα προσεχή έτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Εξ ονόματος του ΑΕΛΚ το λόγο έχει ο κύριος Βέπερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Εάν στρέψουμε τη ματιά μας το 2016, ε, είμαστε πραγματικά επιφυλακτικοί. Η τρομοκρατία, τα προσφυγικά, οι προσφυγικές ροές, η κρίση κλπ. Παρόλα αυτά, ε, την αρχή του χρόνου θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το που είπα και στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Δηλαδή θα ήθελα να αναφέρω επίσης τις επιτυχίες μας, ώστε να ενθαρρύνω τους πολίτες ότι μπορούν, μπορούμε να έχουμε επιτυχίες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδα τις προσπάθειες της Φρεντερίκα Μογκαρίνη ε, και πραγματικά ήμουν υπερήφανος όταν ε, την είδα ε, μαζί με τον πρόεδρο του Ιράν να προχωρά στη συμφωνία, ε, ούτως ώστε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εισφέρει για, την, ε, για το να μην, στο να μην υπάρχουν πλέον πυρηνικά όπλα, πυρηνικό οπλοστάσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. πήραμε επίσης τους αριθμούς του σχεδίου Juncker. Χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ευρώπη υποφελούνται από τα δισεκατομμύρια, από τα κονδύλια τα οποία εμείς αποδεσμεύσαμε. Και η συνδιάσκεψη του κλίματος στο Παρίσι στέφθηκε επίσης με επιτυχία και είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε αυτές τις επιτυχίες το Δεκέμβριο και αυτό είναι το δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω στο επίκεντρο της ομιλίας μου ήταν η συζήτηση με τη Μεγάλη Βρετανία και φαντάζομαι ότι ο Ντέβιτ Κάμερον στο Συμβούλιο ε, παρουσίασε πολλές θετικές προτάσεις και είχε θετική απήχηση. Πολλές από τις ιδέες του Ντέβιτ Κάμερον είναι ιδέες οι οποίες στοχεύουν σε μια βελτίωση της Ευρώπης. Αν υπάρξει μια κοινή προσέγγιση και θέλω να υποστηρίξω τα όσα είπε στο θέμα της ανταγωνιστικότητας για την κοινοτομία, για την καλύτερη ε, ρύθμιση. Ε, εδώ ο Ντέβιτ Κάμερον είχε την πλήρη υποστήριξη, έχει την πλήρη υποστήριξη του ΕΛΚ. Ε, δυσκολότερα είναι τα πράγματα όσον αφορά τις κοινωνικές ε, καταχρήσεις. Ε, ο Ντέβιτ Κάμερ θέλει να καταπολεμήσει αυτά τα θέματα και θα ήθελα να επισημάνω ότι και εμείς στο ΕΛΚ όμως δεν μπορούμε να ανεχτούμε όταν υπάρξουν διακρίσεις εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα, έχω ένα ερώτημα για καταλαβαίνω τις ε, που εκφράστηκαν στο Λονδίνο σε σχέση με την αύξηση των αρμοδιοτήτων στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται κριτικά, με κριτικό πνεύμα. Αλλά εάν δούμε το κείμενο, αναφέρει μια ever closer union of people, ε, μια πιο στενή ένωση ανθρώπων όχι θεσμικών οργάνων. Και αυτή είναι μια πολύ σωστή διατύπωση της ευρωπαϊκής ιδέας. Δηλαδή το να πούμε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έρθουν, οι πολίτες θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά ένας με τον άλλον. Γι' αυτό είμαι υπέρ το κείμενο αυτό ε, να αναγνωστεί ε, προσεκτικά, γιατί πραγματικά μπορούμε να αντιλήσουμε σημαντικά διδάγματα από αυτό το κείμενο. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να φερθώ σε ένα τρίτο θέμα, το μείζον θέμα τη μετανάστευση. Ε, για το ΕΛΚ είναι ξεκάθαρο. Εάν ε, στην ε, Συρία υπάρχει πόλεμος θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ήπειρο αυτό, αυτή. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε, δεν είναι δυνατόν και από την άλλη γνωρίζουμε ότι οι αριθμοί που έχουμε συνιστούν μια τεράστια πρόκληση για μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καθίσω σαφέ για τη δική μου πολιτική ομάδα ότι χαιρετίσουμε το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα πολύ λογικό και όριμο κείμενο. Για μας το ζητούμενο είναι να απεξεργαστούμε το τάχη ταχύτερο ε, τις ε, προτάσεις αυτές ώστε να μπορέσουν να βρουν μια εφαρμογή. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν μιλάμε για 1,1 εκατομμύριο ανθρώπου που έφτασαν στην δική μου πατρίδα, τη Γερμανία, εκατομμύριο χιλιάδες έφτασαν στη Γερμανία και μόνο 40% είναι Σύριοι. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να μεταναστεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να επαναπροωθούν στις πατρίδες τους. Ε, γιατί ξέρουμε τι έγινε στην κολονία την πρωτοχρονιά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο οποίος παραβιάζει το δίκαιο και την παράδοση της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, τον πολιτισμό της Ευρώπης, ο άνθρωπος αυτός τελικά δεν μπορεί να γύρει αξιώσεις, να γίνει δεκτός σε αυτές τις χώρες. Ε, ε, ε, και απευθύνω μια έκκληση στο Συμβούλιο. Αν στο Συμβούλιο δεν πιστωθεί το εξή. Δίνουμε 3 εκατομμύρια στην Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να δώσει αυτά τα χρήματα αλλά τελικά ε, τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν στους αποδέκτες τους και αυτό ζημιώνει ε, τη δική μας υπόλοιψη. Ε, και η συμπεριφορά του Ματέο Ρέντσι ε, συγκεκριμένα πραγματικά ε, ζημιώνει την ευρωπαϊκή αξιοπιστία. δεν θα πρέπει να είμαστε λαϊκιστές, δεν θα πρέπει να δίνουμε ψεύτικες υποσχέσεις. Εμείς θέλουμε να δώσουμε ουσιαστικές απαντήσεις. Κύριε Βέμπερ, η κυρία Γκραπίνη θέλει να σα απευθύνει ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Θα θυμάστε ότι το Δεκέμβριο σας έθεσε ένα παρεμφερές ερώτημα. Συνεχώς μας συμβουλεύετε και συνεχώς λέτε λόγια μεγάλα. Δεν πιστεύετε ότι αυτά που μόλις είπατε τώρα για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ε, δεν θα πρέπει να είναι αυτά που να. Ε, έπρεπε να σκέφτεται η κυρία Μέρκελ εξ αρχής. Μιλάει για τις συνθήκες διατήρησης και προστασίας ε, ε, των αξιών μας και του πολιτισμού μας, αλλά οι συνθήκες αυτές δεν υπάρχουν. Αλλά ήθελα να καλέσω όλου να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της, ε, των προφυσίγων. Και λέω ρητά, εάν στη Συρία, και παρακούστε με, δια, έχουν πεθάνει τόσοι άνθρωποι από τον φίλιο πόλεμο ε, και υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες επειδή ακριβώς γίνονται εκεί οι βομβαρδισμοί. Θα πρέπει ο καθένας να αντιμετωπίσει τις ευθύνε του στην Ευρώπη και εμείς ως Χριστιανική ήπειρο θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να δραπετεύσουν από τον πόλεμο. Και αυτό θα ήθελα να το ακούσουν ειδικά οι Πολωνοί. Δεύτερον, η Ευρώπη έχει κάποια όρια. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε ε, με κάποια νούμερα και θα πρέπει να συζητήσουμε τα... και τις δύο αυτές πλευρές. Εκ μέρους των σοσιαλδημοκρατών έχει το λόγο ο κύριος Σαλόμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου δημιουργήσαν μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση στην πολιτική μου ομάδα. Είναι συναισθήματα τα οποία συνεχώς βιώνουμε μετά τα συμβούλια τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο. Όχι γιατί δεν υιοθετήθηκαν αποφάσεις και δεν επιτεύχθηκαν συμφωνίες. Συνέβησαν αυτά και για τη μετανάστευση και για την ΟΝΕ και για την τρομοκρατία. Το πρόβλημα είναι ότι όταν διαβάζει κανείς τα συμπεράσματα του Ιουνίου, τα συμπεράσματα του Οκτωβρίου τα συμπεράσματα των άτυπων ε, διασκέψεων του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου πρέπει να διαβάσει πολύ προσεκτικά για να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι τα ίδια συμπεράσματα. Είμαστε καταδικασμένοι για άλλη μια φορά να ακολουθούμε την ίδια αλληλουχία. Η Κομισιόν προετοιμάζει και προτείνει, τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο υιοθετούν αποφάσει, αλλά μετά όταν πάνε στι πρωτεύουσε του αγνοούν και δεν ε, εφαρμόζουν ολοκληρωτικά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στα συμβούλια. Αυτός είναι ο συσήφιος μύθος. Συνεχώ επιστρέφουμε στην αρχή. Ας μιλήσουμε για τα θέματα. Τρομοκρατία παραμένει άλυτο το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών. Σήμερα το πρωί ο κύριος Γιούνκερ μας επισήμανε ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση με αυτή του 2001 μετά τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη. Είναι αληθές ότι επικροτώ την πρόταση που ανακοίνωσε ο κύριος Γιούνκερ σήμερα το πρωί για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μετανάστευση. Δεν λειτουργούν τα hot spot δεν λειτουργεί η επανεγκατάσταση ή μετεγκατάσταση και επιδεινώνεται το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό κλίμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομία απουσιάζει από τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου, αλλά η ανεργία παραμένει σε ψηλά επίπεδα, οι ανισότητες οξύνονται και η έλλειψη ευκαιριών επικρατεί. Θα δεχθούμε να είμαστε σαν το σύσυφο, δηλαδή καταδικασμένοι να ξαναγυρνάμε από την αρχή. Ας ακούσουμε τον τόνο τον οποίο παραθέσατε εσείς πρόεδρε Τούσκ. Ας αποφύγουμε τη δική μας αυτοκτονία. Αν δεν την αποφύγουμε θα ολοκληρωθεί ο μύθος του Σισύφου με εμάς τους ιδίους. Θα είμαστε ανίκανοι να προχωρήσουμε και αυτό θα σημάνει τον πολιτικό μας θάνατο. Ο κύριος Βανόρντεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να ασχολείται περισσότερο με το να βρει κάποιο ρόλο η ίδια για να διατηρήσει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και τελικά δεν κάνει τίποτα ή μάλλον επιδεινώνει τελικά τα πράγματα. Πολλά από τα προβλήματα που έχουμε, οικονομικά, πολιτικά, προβλήματα ασφαλεία, είναι συνέπεια τη ίδια τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρετίζουμε την υποστήριξη κρατών μελών και κάποιων ε, λογικών ευρωβουλευτών που θέλουν να προωθήσουν τι μεταρρυθμίσει που ζητά ο Ντέβιτ Κάμερον. Νομίζω ότι θα πρέπει με ενθουσιασμό να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι ε, αιτήσει που κάνει ο Κάμερον για μεταρρυθμίσει και αλλαγέ. Θα πρέπει οι ευρωβουλευτέ να συνειδητοποιήσουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν θέλουν όλο και στενότερη ένωση, θέλουν υπεύθυνε κυβερνήσει, υπεύθυνε για τι δράσει του. Θέλουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα κοστίζει λιγότερο, μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποτελεσματική στη δαπάνηση των πόρων, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μειώσει τη γραφειοκρατία, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καταρρύψει τα εμπόδια στο εμπόριο και στην ανταγωνιστικότητα, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πολύ γρήγορα θα συνάψει εμπορικέ συμφωνίε με χώρε όπω η Ινδία ή που θα καταφέρει να ολοκληρώσει το TTIP. Δεν θέλουν οι πολίτες να τροποποιηθεί η ζωή τους από την μαζική αυτή έλευση προσφύγων από άλλες χώρες και προφανώς οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να υπάρχει καλύτερη ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Είναι πολύ λογική τελικά η πολιτική του David Cameron απέναντι στους πρόσφυγες αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αιτία του προβλέματος, βοηθά τους ανθρώπους που βρίσκονται σε, προ... καταβλισμούς και προσπαθεί να βοηθήσει τις πιο ευάλωτες ομάδες. Ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μειώσει τα να καταπολεμήσει τα πραγματικά αίτια καθώς επίσης και τις, να εφαρμόσει τις διεθνείς συμφωνίες που υπάρχουν όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης. Και όπως υπόθηκε, οι περισσότεροι μετανάστες δεν έρχονται τελικά από τη Συρία. Η τρομοκρατία είναι ξεχωριστό ζήτημα, αλλά συνδέεται με τη μετανάστευση. Είμαστε υπέρ της συμφωνίας για τα PNR, σημαντική πρόοδο εκεί, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ακόμα περισσότερη πρόοδο. Η μεγαλύτερη συνεργασία που θέλουμε θα επιτευχθεί καλύτερα μεταξύ των εθνικών διοκτικών αρχών, των εθνικών σωμάτων την αστυνομία. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι φιλελεύθεροι έχουν το λόγο. Ο πρόεδρος τους, κύριος Φέρφορστατ. Κύριε Πρόεδρε, ε, δίστασα να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση γιατί πραγματικά επαναλαμβάνουμε συνεχώς αυτά τα οποία έχουμε πει. Νομίζω είναι η τέταρτη πέμπτη φορά που έχουμε ακριβώς την ίδια συζήτηση και συμφωνώ με τον κύριο Γκερέρο πραγματικά χρησιμοποίησε μια πολύ ακριβή μεταφορά, το μύθο του Σισίφου. Κάθε φορά λέμε χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή. Πού είναι. Εδώ και μήνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε στο τραπέζι του Συμβουλίου αυτή την πρόταση και ακόμα την αναμένουμε. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα να παρακολουθήσουμε και να εξασφαλίσουμε τα εξωτερικά μα σύνορα. Και όταν ακούω, κύριε Βανόρντο, να επενείται την πολιτική του κυρίου Κάμερον για του πρόσφυγε, Σω ε, ε, ε, Ίσως πάτε μαζί μου και με άλλους εθελοντές στα στρατόπεδα, στο Καλέ και στη Δουμκέρκη που ζουν μέσα στη λάσπη παιδιά τα οποία δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι η λεγόμενη ανοιχτή πολιτική μιας συντηρητικής κυβέρνηση Πραγματικά είναι όνειδος αν μεταβείτε εκεί και, δείτε σε τι συνθήκες διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι εύκολο να μιλάει κανείς για τα νότια σύνορα της Ευρώπης εάν διαπιστώνει τι συμβαίνει στα δυτικά σύνορα της Ευρώπης και ο δικός μου φόβος είναι ότι τελικά δεν εφαρμόζεται πλέον το Σέγγεν στη Δανία, στη Σουηδία, στην Αυστρία, στη Σλοβενία, στην Ουγγαρία. Ε, και τι θα συμβεί αν κάνει το ίδιο και η Γερμανία μεθαύριο. Αυτό θα μπορούσε να είναι το τέλος του Σέγγεν, το τέλος της Ευρωπαϊκής. Ωραία, ωραία. Αυτό ακριβώς θέλετε. Θέλετε να επιστρέψετε στη Βρετανική σας αυτοκρατορία, η οποία δεν υφίσταται πλέον. Αλλά η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα όλα αυτά καταραίουν λόγω έλλειψης αποφασιστικότητας εκ μέρους των χωρών μελών. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή στην οποία λείπει η αποφασιστικότητα, αλλά το Συμβούλιο. Και ελπίζω κάθε φορά που πρόκειται να ληφθούν αποφάσει για την ευρωπαϊκή συνοριοφαλική, σε νέα νέα μεταναστευτική πολιτική, σε ένα σύστημα χορήγηση ε, ασύλου, ε, η ε, πανεγκατάσταση των προσφύγων, ένα νέο σύστημα προτάθηκαν 160, προτάθηκε ο αριθμός των 160.000 ε, και τελικά μόνο 290 τελικά μπόρεσαν να εγκατασταθούν κανονικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο σύστημα. Ε, κύριε Τούσκα, ε, θα έχετε μια έκτατη σύνοδο κορυφής στις 18 Φεβρουαρίου στο Brexit. Ε, κάνετε μια έκτακτη σύνοδο και ε, για, την, ε, για το θέμα των προσφύγων. Νομίζω το θέμα του Brexit μπορεί να περιμένει. Νομίζω ότι το πιο επίγον θέμα είναι το ζήτημα της εγκατάστασης των προσφύγων, ένα νέο σύστημα χορήγησης ασύλου και ε, το ζήτημα της ονοριοφυλακής. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο σημαντικά από τα ζητήματα του Brexit. Γιατί ενδεχομένως ε, η Μεγάλη Βρετανία ε, θα παραμείνει εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εάν δεν επιλύσουμε το ζήτημα των προσφύγων, τελικά θα καταρρεύσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Φέρχοφστατ, έχετε ε, την επιλογή να δεχτείτε ε, ερωτήσεις που σας απευθύνονται. Ε, ολόκληρο, ομάδα ο ΚΙΠ. Αλλά θα τους πάρουμε τη σειρά. Ο πρώτος ήταν ο κύριος Πάτον. Κύριε Φερχόφστατ, εσείς και εγώ ερχόμαστε από τελείως διαφορετικά μετερίζια. Πάντοτε μου αρέσει να σας ακούω και σέβομαι αυτά που λέτε, γιατί σε αυτά που λέτε φαίνεται μια σαφή, ξεκάθαρη και λογική πολιτική. Απλά είναι εντελώς αντίθετη από τη δική μου. Πράγματι πιστεύετε στην καλύτερη ενσωμάτωση, καλύτερη ένταξη. Ξέρετε το πραγματικό νόημα της μιας πιο στενής Ευρώπης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό και εγώ το σέβομαι. Δεν σέβομαι συμπατριώτες μου που δεν το γνωρίζουν. Να σας ρωτήσω το εξή: Όταν έχουμε το δημοψήφισμα στη Βρετανία, μπορείτε να έρθετε να επιχειρηματολογήσετε για την παραμονή μας, έτσι ώστε να έχουμε μια σαφή και έντιμη συζήτηση. Ο κύριος Φερχόφστατ, παρακαλώ. Δέχομαι την πρόσκληση. Νομίζω ότι ο πρώτος που γελάει είναι ο κύριος Φάρατζ. Του αρέσει να γίνεται συζήτηση γι' αυτό. Αλλά πρέπει να προχωρήσετε το συλλογισμό σας. Ποια η κατάσταση θα είναι, σε ποια κατάσταση θα είναι η Βρετανική οικονομία χωρί την εσωτερική αγορά της Ένωσης. Ποιο θα είναι το βάρος της, του City του Λονδίνου, αν δεν μπορεί να συνελάσσεται σε ευρώ, όπου το 70% και το 80% του trading στο City του Λονδίνου γίνεται σε ευρώ. Νομίζω ότι η Βρετανία πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη και είναι εντελώ τρελό να νομίζει κανεί ότι μπορεί να πάει πίσω στην ιστορία και να τα κάνει όλα μόνο του. Δεν δουλεύουν αυτά τα πράγματα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία του σήμερα. Το ρόλο έχει τώρα η κυρία Τσούμπερ για την Ενωμένη Αριστερά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούσαμε πώς πρόκειται να αποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσφυγική κρίση. Και είδαμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά επιθυμεί να καταφέρει να ενδυναμώσει κάποιους ήδη φυστάμενους μηχανισμούς. Και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι θέλει να απορρίψει οποιονδήποτε δεν θα μπορεί να πάρει άσυλο ή να καλυφθεί από το καθεστώς διεθνούς προστασίας βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υποστηρίξει την Ελλάδα και την Ιταλία κυρίως για τις επιχειρήσεις επιστροφής, Ψαστικά είναι επιχειρήσεις έκδοσης, απέλασης. Τρία δισεκατομμύρια στην Τουρκία προκειμένου οι πρόσφυγες να μείνουν εκεί. Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια αξιοπρέπεια κανείς δεν γνωρίζει. Το πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε η ίδια μία κατάσταση και διονύζει μία κατάσταση επεμβαίνοντας στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι θα έπρεπε η Frontex και η Ευρωπόλ πέρα από τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, να είναι σε θέση πραγματικά να βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τεράστια ανάγκη βοήθειας και υποστήριξης αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δημιουργηθούν ασφαλείς, νόμιμες οδοί, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη χάνουν ανθρωπιστικής προστασίας. λόγο κυρία Τσεκ, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, στα θεωρία. Η συνάντηση κορυφής τον Δεκέμβριο άσκησε κριτική στις κυβερνήσεις ότι δεν επιλύθηκε το ζήτημα των προσφύγων. Και αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα για μια βελτίωση της πολιτικής. Ωστόσο αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ένα μήνα μετά είναι ότι η διαχείριση της κρίσης στο θέμα των προσφύγων ε, δεν έφερε αποτελέσματα. Τα hot spots ε, δεν λειτουργούν. Η κατανομή των ετούντων άσυλο δεν λειτουργεί. Ε, και όπως είπαμε 290 είναι αυτοί οι οποίοι εγκαταστάθηκαν επιτυχώς από τους 160.000. Ε, είναι δυνατόν με αυτά τα δεδομένα να πιστέψει ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ότι ε, οι ευρωπαίοι πολιτικοί μπορούν να βρουν ε, λύσεις. Κύριε Τούσκ, ελπίζω η επόμενη συνάντηση κορυφής να είναι πιο ουσιαστική. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να εξαθεί με τις Βρυξέλλες. Η Ευρώπη είναι οι χώρες μέλη. Ε, τι θα γίνει εάν ε, επανα... ξαναφτιαχθούν τα σύνορα στο Σέγγεν. Ε, αυτό συνιστά μία πισθοδρόμηση και θα πρέπει να επικρίνω και την κυβέρνηση της Αυστρίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι κοινικός απέναντι στους πρόσφυγες. Λέει όσο περισσότερα σύνορα τόσο μεγαλύτερη πίεση στην Ελλάδα, άρα τόσο γρηγορότερα θα βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση. Αλλά αυτό είναι απόλυτος ε, κινησμός θα πρέπει να βρούμε μία λύση και όπως ε, υπόθηκε σωστά το Brexit μπορεί να περιμένει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λούνετσε και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Φάραντ. Ευχαριστώ. Με χαρά θα καλωσορίσω τον κύριο Φερχόφστατ στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υπερασπιστεί την παραμονή της Βρετανίας στην Ένωση. Έχει γίνει ειλικρινή συζήτηση και θα χαρούν πάρα πολύ οι φιλελεύθεροι να συζητήσουν μαζί μας για αυτό το θέμα. Έχει περάσει ένας μήνας από το τελευταίο Συμβούλιο και έχουν γίνει κοσμογονικές αλλαγές εν μεταξύ. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος, έχει καταλάβει την τρέλα των Ευρωπαίων ηγετών, το σχέδιο Juncker, το κάλεσμα της Μέρκελ, διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές κουλτούρες χωρίς ελέγχους ασφαλείας απειλούν τη συνοχή των κοινωνιών μας και κακοποιούνται επειδή το λένε όσοι το λένε αυτό και το περιγράφουν. Στο Μόναχο, ο σιδηροδρομικός σταθμός έκλεισε λόγω τρομοκρατικής απειλής. Ήρθαν πληροφορίες από τη Συρία και το Ιράκ. Στον ίδιο σιδηροδρομικό σταθμό, το Σεπτέμβριο υπήρχε κόσμος που είχε πλακάτα ε, πρόσφυγες καλωσορίσατε. Δι, φαίνεται τι σημαίνει όλο αυτό. Στην κολονία επίσης το είδαμε. Χίλιοι άνδρες στο δρόμο επιτέθηκαν σεξουαλικά και παρενόχλησαν γυναίκες. Είναι από τα πιο επονίδιστα γεγονότα συμβάντα κατάλυσης της δημοσίας τάξης. Παρόλα αυτά, ο τύπος και η αστυνομία προσπάθησαν να το καπαρώσουν, να το καλύψουν κάπως και Ορισμένοι δημοσιογράφοι είπαν ότι οι νέες, νεαρές Γερμανίδες πρέπει να αλλάξουν και την ενδυμασία τους όταν κυκλοφορούν στους γερμανικούς δρόμους, κάτι το οποίο είναι εξόφθαρμη προσβολή για μένα. Όλα αυτά έχουν γίνει κοινό τόπος μέρος της καθημερινότητάς μας και πρέπει να στείλουμε το μήνυμα και να πούμε ότι αυτές οι επιθέσεις ποτέ δεν μπορούν να είναι αποδεκτές σε καμία ευρωπαϊκή πόλη, μικρή ή μεγάλη και θα κάνουμε το παν για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα στην επόμενη σύνοδο ο κύριος Κάμερον θα θέλει να ξεκινήσει την επαναδιαπραγμάτευση και σίγουρα θα υπάρξει ε, ε, συμψηφισμός και θα υπάρξει συμβιβασμός ε, στα ίσονος σημασία ζητήματα και θα επιστρέψει από τη Σύνοδο με ένα χαρτί πολλά υποσχόμενο για τη σχέση της Βρετανίας με την Ένωση, αλλά δεν θα μιλήσει καθόλου για τη δυνατότητά μας να ανακτήσουμε τον έλεγχο των συνόρων μας. Και οι Βρετανοί γνωρίζουν ότι σε λίγα χρόνια οι, όσοι διέπραξαν αυτά τα δικήματα στην κολονία και στο σταθμό του τρένου θα έχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο και θα μπορούν να έρθουν στη Βρετανία. Ε, ο σχολιαστής, η, η σχολιάστρια Άλεξον Πίρσον της Daily Common είπε ότι μετά την κολονία το δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με την ασφάλεια των ε, Βρετανίδων γυναικών. Πρέπει να πολεμήσουμε για το δικαίωμα των κορών μας και των εγγονών μας να ζήσουν όπως θέλουν, να χαμογελούν και να ντύνονται όπως θέλουν στο δρόμο. Και ας τους δώσουμε να καταλάβουν επιτέλους. Το 2016 θα είναι η χρονιά που θα φέρουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας παρακαλέσω το εξή. Ε, ε, υπήρξε μια ερώτηση προς την κυρία Λούνετσεκ. Δεν ε, την πρόσεξα, αλλά καταρχήν θα, να πάρει το λόγο ο κ. Φερφχοφστάτ για τον κύριο Φάραξ να πω ότι η σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση είναι φαινόμενα που υπάρχουν και στη Βρετανία και είναι και βρετανική ορολογία ούτως ή άλλως, την οποία ε, χρησιμοποίησαμε οι υπόλοιποι ε, χώρες και οι υπόλοιποι λαοί. So, Is this reasonable We've had it more than from this gentleman. Είναι λογικό, λέει ο κύριος Φάρ, να δεχόμαστε αυτές τις προσβολές. Σίγουρα είμαστε όλοι ισότιμοι, αλλά απαιτούμε αξιοπρέπεια και σεβασμό. Δεν μου δώσατε την ε, ευκαιρία να πω τίποτα, κύριε Φάραντζ. Εσύ με την αποτελεσματικότητα που σας διακρίνει, βιαστήκατε να πάρετε το λόγο, κύριε Φάραντζ. Ο κύριος ε, ε, Φέρχοφστ αναφέρθηκε σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε σχέση με το κόμμα, με το κόμμα του κυρίου Φάρατζ. Ε, παρακαλείται να τις ε, αποσύρει. Κυρία Στόρχ, θέλατε να θέσετε μία ερώτηση προς την κυρία Λούνατσεκ. Μάλιστα κύριε Σούλτσεκ. Κυρία Λούνατσεκ, μια σύντομη ερώτηση. Μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας, πότε έχετε την... Ε, μετά από ποιο αριθμό ε, προσφύγων σε αριθμού σε εκατομμύρια ε, θα πρέπει η Γερμανία να προστατεύσει τα σύνορά της. Ε, απάντηση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η ερώτηση αυτή δεν μπορεί να απαντηθεί με συγκεκριμένου αριθμού, με νούμερα. Τι θα κάνατε εσεί εάν εσείς κάτι που δεν ελπίζω είσαστε στην κυβέρνηση και λέτε ότι ε, η Γερμανία θα δεχτεί ένα εκατομμύριο ε, και μετά έρθει ο εκατομμυριστός πρώτος. Τι θα κάνετε, θα το στείλετε πίσω. Το λόγο έχει τώρα ε, η κυρία Μάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2015 ομοιάζουν τελικά με συμπεράσματα από προηγούμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Η μόνη λύση όμως η οποία θα μπορούσε να προταθεί είναι το κλείσιμο των συνόρων, κάτι το οποίο όμως δεν θέλουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά στην πράξη το κάνουν πολλές χώρες. Αρκεί να δείτε λίγο τις ειδήσει τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι ετούντες άσυλο, αρκεί να δούμε τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2016. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσει σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, οι κάτω χώρες κτλ. Επίσης έχουμε τρομοκρατικές επιθέσεις, πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε σεξουαλικές παρανοχλήσεις στο Ντόρτμουθ, στο Καλέ ένας ε, Ολλανδός ε, βουλευτής έπεσε και αυτός θύμα επιθέσεων. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον για τις κάτω χώρες, να κλείσουμε τα σύνορά μας. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προασπίσουμε τον πολιτισμό μας και την ευημερία μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκχωρήσεις στα ζητήματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Ζαριανόπουλος. αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. της ΟΝΕ δηλαδή ενιαία εφαρμογή της αντεργατικής πολιτικής για τα κέρδη του κεφαλαίου συμβούλια ανταγωνιστικότητας και δημοσιονομικά συμβούλια για αυτόματη περικοπή μισθών συντάξεων και κοινωνικών παροχών ενοποίηση των αγορών. αυτά συμπληρώνονται με κλιμάκωση των εμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων με πρόσχημα και την αντιτρομοκρατική εκστρατεία για κατάκτηση νέων αγορών πηγών και δρόμων ενέργειας. αυτά γεννάνε ανεργία φτώχεια πολέμους το προσφυγικό δράμα το συμβούλιο αποφάσισε ένταση καταστολής κατά προσφύγων και μεταναστών hot spot διαλογής πάνθηνου εργατικού δυναμικού που θα περνά τα έξυπνα σύνορα ενώ η πλειοψηφία θα αναχαιτίζεται ή θα πνίγεται στο αιγαίο θα απελάβνεται ή θα αποθηκεύεται στην ελλάδα. η δημιουργία κατασταλτικής ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής με δικαίωμα επέμβασης χωρίς τη συνένεση των κρατών βάζει στη λιμιτόμο των ευρωενωσιακών συμφερόντων τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελλάδας προωθεί παζάρια στη διαχείριση του αιγαίου με την τουρκία υπό ευρωανατολική ομπρέλα. αποδεικνύεται καθημερινά η ευρωπαϊκή ένωση του Καπιταλισμού που υπηρετεί δεν αλλάζει. μόνο η πάλη των λαών μπορεί να ανατρέψει ριζικά αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Θέλετε να το λόγο επί διαδικαστικού, κύριε Φέρχοφστατ. θέσετε μια ερώτηση και σας απάντησα ότι αν πάτε στο Google και βάλετε harassment, ε, σεξουαλική παρενόχληση, θα έχετε την απάντηση που επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση, λέει ο κ. Σούλτς. Το λόγο τώρα εκ μέρου του ΕΛΚ, ο κ. Ε, Λαμασούρ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Α είμαστε έντιμοι όσον αφορά το θέμα των προσφύγων. Όλοι έχουμε αποτύχει. Οι χώρε μέλη καταρχήν τόσο πιο μεγάλες όσο και πιο μικρές, οι πιο ανοιχτέ όσο και οι πιο κλειστές. Οι χώρες εκτός του Σέγγεν καθώς και οι χώρες εντός ε, Σέγγεν και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, πρόβλημα, ε, το πρόγραμμα της επανεγκατάστασης των προσφύγων δεν αφορούσε παρά μόνο 10% ε, των πραγματικών εισόδων και όπως υπόθηκε εφαρμόστηκε μόνο κατά ένα ή δύο της χιλίης. Το δύο μπορούμε να αντλήσουμε είναι ξεκάθαρο οι εθνικοί εγωισμοί δεν οδηγούν πουθενά. Δεν πρόκειται πλέον για μια δυνατότητα αναλλακτική λύση. Μια χώρα μέλος ε, δεν μπορεί να ρίχνει το πρόβλημα ε, στους γείτονές της το πρόβλημα και από την άλλη να στρέφεται σε αυτούς για να ζητήσει χρηματοδότηση. Δεν μπορεί μια χώρα μέλος να αποφασίζει μόνη να υποδεχτεί όλους όσους θα εμφανιστούν και στη συνέχεια να ζητάει βοήθεια σε εκείνους τους εταίρους που έχουν διαφορετικές πολιτικές επιλογές. Ποια από τις χώρες ε, μέλη μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη το πρόβλημα σε μια χώρα προέλευσης ε, που βρίσκεται σε πόλεμο ή σε μια χώρα διέλευσης όπως είναι η Τουρκία ή η Λιβύη. Η λιβυη οσον αφορά δε το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πώς, μπορούμε, πώς μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι μια κυρίαρχη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αφήνει τις χώρες ε, μέλη να περηφανεύονται ότι δεν εφαρμόζονται τις ίδιες τις αποφάσεις. Ε, Ας δούμε κατάματα την ε, πραγματικότητα. Μόνο ενωμένοι ε, μπορούμε να κυριαρχήσουμε στα προβλήματα. Υπάρχει ένας ε, χρόνος για το συνέστημα και υπάρχει και ένας χρόνος για την λογική. Επίσης υπάρχει ένας κατάλληλος χρόνος για να αναλάβουμε την ευθύνη που μας προσήκει. Η κυρία Φαγιόν έχει το λόγο δύο λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μετά το Συμβούλιο δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξη όταν μιλούμε για μετανάστες και πρόσφυγες γιατί παντού υπάρχουν προβλήματα στην ε, υποδοχή, στην εγκατάσταση, στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με, ε, την Τουρκία και ενώ προσπαθούμε να ρίξουμε τα σειρματοπλέγματα, να διονται νέα σειρματοπλέγματα και οι άνθρωποι είναι όλο και λιγότερο ανεκτικοί, γιατί ανησυχούν. Ανησυχούν ότι δεν υπάρχει πια η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Ανησυχούμε για το τι θα γίνει την Άνοιξη όταν έρθουν ακόμη περισσότεροι πρόσφυγες προς την Ευρώπη. Πριν από μερικές μόλις μέρες Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από μερικά χρόνια, πριν από τρία χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνη. Αυτό θα έπρεπε να είναι το κίνητρό μα για περισσότερη συνεργασία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κανένα κράτο ε, να αντιμετωπίσει, γιατί δεν μπορεί κανένα κράτος να αντιμετωπίσει μόνο την ε, μεγάλη αυτή πρόκληση. Πρέπει να συνεργαστούμε για κοινά αποτελέσματα. Πρέπει να συνεργαστούμε, να αφήσουμε κατά μέρο τους εγωισμούς, τους εθνικισμούς, τις ακρότητες. Ίσως θα ήταν καλύτερο να σταματήσουμε και να συνομιλούμε, να, να δίνουμε τόσο πολύ βάρος στις συνομιλίες και να κοιτάξουμε να δράσουμε περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν ύστερα από εβδομάδες που συζητούμε το θέμα να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και να μην γίνεται τίποτα. Μπορεί να μετατραπεί αυτό στην πολιτική μας αυτοκτονία. Αν δεν πράξουμε τίποτα δεν θα πλέον, ε, δεν θα έχει καν λόγο ύπαρξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Φωτσίγα. Πρόεδρε, το Συμβούλιο θα πρέπει να αναζητήσει όρους ώστε να περιγράψει το συσχετισμό μεταξύ της τρομοκρατικής απειλής και της μεταναστευτικής ε, πολιτικής. Πρέπει να κοιτάξουμε να καταπολεμήσουμε αυτούς που δοξάζουν την τρομοκρατική απειλή. Φιρυπίν, παλαιστινιακή πλευρά. Και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε τις σχέσεις μεταξύ ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όλο και πιο έντονος ο κίνδυνος του Brexit και έχει έρθει η ώρα να τα συστήσουμε αυτά. Στη συνέχεια Κονζάλε Πένιας. Ευχαριστώ. Τη εβδομάδα αυτή ολοκληρώνεται ένα εξάμεινο, ευρωπαϊκό εξάμεινο, με την ε, μεγάλη επίθεση αυτή που έχει γίνει σε βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε με ένα μνημόνιο που είναι ό,τι χειρότερο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Δεν θέλουμε την Ευρώπη των κοινωνικών περικοπών. Θέλουμε το κράτος ευημερία και θέλουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να προχωρήσει προς τα κοινωνικά δικαιώματα. Έχουμε μια πιο άνηση Ευρώπη όσο περνάει ο καιρός και δεν μιλάμε γι' αυτό, για τις δύο ταχύτητες που χωρίζουν την Ευρώπη του Νότου από την υπόλοιπη, του Νότου που δεν έχει δικαιώματα κοινωνικά καθόλου. Και τι η ηθική δύναμη μπορεί να έχει ο πρόεδρος της Επιτροπής που εκπροσωπεί πολυεθνικές και μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Κύριε Γιούνκερ, η Ευρώπη πρέπει να δίνει απαντήσεις στην ανθρωπιστική κρίση. Όχι να δίνουμε χρήματα για να κάνουμε ακόμα πιο αδιάβατα τα σύνορα, αλλά να βοηθάμε στην ανθρωπιστική κρίση. Φεράρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο διχασμός, η έλλειψη εμπιστοσύνη χαρακτηρίζουν τις ευρωπαϊκές χώρες για θέματα όπως είναι Οικονομική και Νοσματική Ένωση, μετανάστευση και ασφάλεια. Σήμερα ακόμα ο πρόεδρος Γιούνκερ μας μίλησε για πολλαπλές κρίσεις, λέγοντας ότι κάποιοι επικρίνουν πολύ εύκολα τις Βρυξέλλες αντί να κοιτάξουν να δουν τι γίνεται στις δικές τους χώρες. Κύριε Γιούνκερ, Αναφέρεστε στην Ιταλική κυβέρνηση μήπως, γιατί διαβάζοντας τον τύπο σήμερα είδαμε ότι σας εκνεύρισε η συμπεριφορά του κύριου Ρέντσι. Και θεωρείτε τη συμπεριφορά αυτή ότι δείχνει ότι δεν είναι κατάλληλος νομιλητής για τις Βρυξέλλες. Εμείς δεν εκπλησόμεθα. Εδώ και καιρό καταγγέλουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει καν εκλεγεί από τους πολίτες. Δεν μπορεί μια τέτοια κυβέρνηση να αντιπροσωπεύει τους πολίτες και τις ανάγκες τους σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα το κατάλαβε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έλλειψη διαλόγου ανάμεσα σε εσά και τον Πρωθυπουργό μας ε, Ρέντσι είναι επίσης ένα στοιχείο. Αλλά όχι μόνο, εδώ δεν υπάρχει διάλογος με τους πολίτες, οι οποίοι έχουν κουραστεί γιατί τους επιβάλλεται πολιτικές που τους αδικούν. Υπάρχει μια πραγματική κρίση αντιπροσώπευσης λοιπόν. Εφόσον υπάρχουν τέτοιες διαφορές, τέτοια επιφύλαξη και τέτοια έλλειψη κατανόησης, μετά από τόσες θεσμικές <coughs> συναντήσεις και λοιπά εγκρίνονται μέτρα και κλεισμένων των θυρών, γιατί στην συνεδριάσεις κομισιών γίνονται και κλεισμένων των θυρών, δεν υπάρχουν πρακτικά. Δεν γνωρίζουμε τις θέσεις των διαφόρων χωρών μελών. Μπροστά σε όλα αυτά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να βασιστεί καλύτερα σε μια άμεση δημοκρατία, κάτι το οποίο όμως δεν γίνεται και δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει τελικά. Και κυρίως πώς προστατεύονται τα συμφέροντά μας. Πρόεδρε Γιούνκερ, πρόεδρε Τούσκ, εξηγήστε μας καλύτερα. Εξηγήστε μας πού έχουν φτάσει τα πράγματα. Θα ήθελα να έχω μια απάντηση συγκεκριμένη γι' αυτό. Ευχαριστώ. Merci, κυρία Μπιτσότο για ένα λεπτό. Συνάδελφοι, είμαι σε σύγχυση και δεν καταλαβαίνω καθόλου τι γίνεται. Ανησυχώ, διότι πριν από λίγου μήνε εδώ πέρα λέγαμε ότι η μετανάστευση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη. Τώρα, ε, πολύ δειλά, αρχίζουμε να λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα. Και ενώ συνεχίζουμε να συζητάμε τι δυσκολίε, τελικά βλέπουμε ότι έχουμε γονατίσει από τι υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει. Μόλι πέρσι έφτασαν ένα εκατομμύριο πρόσφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι ροέ συνεχίζουν να διωγγώνονται. Και εντωμεταξύ με τι αποφάσει σα έχετε φέρει την Ευρώπη σε χάο. Οι πόλει μα έχουν κατακλειστεί από ε, χιλιάδε μετανάστε που ε, εκμεταλλεύονται τη φιλοξενία μα και ε, βιάζουν, ε, κλέβουν υπάρχοντα και εκμεταλλεύονται το σύστημα. τα επεισόδια στην κολονία δείχνουν ότι το ευρωπαϊκό σύστημα δεν λειτουργεί. Ή κλείστε τα σύνορα ή βοηθήστε πραγματικά τους πολίτες βοηθώντας, αξιοποιώντας τους πόρους και όχι τους ε, υποτιθέμενους πρόσφυγες. Προστατεύστε τις πόλεις μας και κοιτάξτε να σταθεροποιήσετε τις χώρες προέλευσης. Χρειάζονται πολύ λίγοι κανόνες και φτάνουν τα μπλα μπλα που μόνο προβλήματα μας δημιουργούν. Είναι συναντηνός για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, όταν η επιτροπή ανακοινώνει μεγαλεπίβολα σχέδια για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και της τρομοκρατίας επιβεβαιώνομαι ότι πρέπει να αλλάξουμε επιτρόπους του συμβούλους αυτών και τους δυο. τσιγαντιστέ σκοτώνουν αθώους και αποφασίσατε να χαρίσετε 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην τουρκία η οποία βοηθά εξοπλίζει και συνδιαλέγεται με το ισλαμικό κράτος. σας καλώ λοιπόν να δεχτείτε την τουρκία στην ένωση και αντίστοιχα σφίγγει η ελλάδα να λυθούν τότε αυτόματα όλα τα προβλήματά σας. πού είναι το σχέδιο επανεγκατάσταση και αναδιανομή το σχέδιο επανεισδοχής. τώρα μας λένε ότι θα δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό σώμα συνοριοφυλάκων και ακτοφυλακής. κύριοι της επιτροπής απαλλάξτε μας από την υποχρέωση να ακούμε τις ανοησίες σας. πόσος χρόνος και χρήμα θα χρειαστούν για να τις καταστήσετε επιχειρησιακά έτοιμες; βάσει ποιά συνθήκη και νομοθεσίας θα επιχειρούν; από πού θα βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια; λάβατε υπόψη σας αρχές της αναλογικότητα και τη επικούρικότητα. η συνθήκη της ένωσης ορίζει ρητά ότι η φύλαξη των εθνικών συνόρων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών στην ιταλία σχεδιάζεται την εμπλοκή τη ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη μεσογείου μια δύναμη η οποία κάλλιστα με την άδεια και το συντονισμό τη ελλάδο μπορεί να επιχειρεί και στο αιγαίο. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κύριο Γκονζάλε. Πόντ Πόντς για 1,5 λεπτό τώρα. Ευχαριστώ. Ξεκινάει μια δύσκολη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το ξέρουμε ευθύ εξ αρχή. Τα παλιά προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, όπω έλεγε και ο Ρίκε Γκερέρο. Μερικά όμω με νέο πρόσωπο, όπως η επίθεση εκείνη εναντίον γυναικών στο κέντρο της Ευρώπης, η ξενοφοβία. Έχουμε όμως και νέα προβλήματα, όπως είναι η διαδικασία κατά της Πολωνίας που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Τάσκα, πρόεδρος του Συμβουλίου, θα μπορούσε να παρουσιάσει τη θέση του Συμβουλίου. Τον ακούσαμε βέβαια πριν, ακούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαι μάντη, αλλά μπορώ να πω ότι την επόμενη χρονιά θα εξακολουθούμε να μιλάμε για τη μετανάστευση, γιατί δεν τέλειωσε ο πόλεμο στη Συρία, γιατί μετά το χειμώνα θα έρθουν νέα κύματα προσφύγων, γιατί χώρε μέλη δεν εφαρμόζουν μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση δεν είμαι μάντη, αλλά θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τη τρομοκρατία, γιατί εξακολουθεί να είναι άμεση απειλή και δεν μοιραζόμαστε τις πληροφορίε που έχουμε, δεν τι ανταλλάσσουμε. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Υπάρχουν και οι νέοι ε, πολίτες, τα νέα θύματα, οι Γερμανοί στην Τουρκία για παράδειγμα μετά από την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση εκεί. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την ενιαία αγορά, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την Κίνα. Δεν είμαι μάντη, λέω, αλλά θα συνεχίσουμε να μιλάμε και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί η Ευρώπη χωρί Ηνωμένο Βασίλειο χάνει. Αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο χωρί Ευρώπη επίση χάνει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να το πούμε στου Βρετανού φίλου, όπω και εκείνοι το λέγανε στου Σκοτσέζου. Ευχαριστούμε κύριε Γκονζάλες. Υπάρχει μπλε κάρτα για σά. Δέχεστε. Κύριε Κοζάλες, με ακούτε. Δέχεστε μπλε κάρτα. Παρακαλώ, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχει καθοριστική σημασία και το να καταλήξουμε στο ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική για την προσβυγική κρίση μεταξύ της Ισπανίας και της Ελλάδας. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καταλήγουμε σε αυθαίρετες αποφάσεις, κατά αποκοπή λύση, αλλά να κοιτούμε πού μπορεί καλύτερα να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική. Μήπως έχετε κάποιες ιδέες να προσφέρετε. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της όσον αφορά τους πρόσφυγες και το κάνει. Είναι πολύ σημαντικό το Συμβούλιο να πάρει στα σοβαρά τις ανάγκες των Ευρωπαίων και ελπίζω να το κάνει. Αλλά κυρίως είναι πολύ σημαντικό οι χώρες μέλη να εφαρμόζουν τόσα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν το κάνουν. Η κυρία Ροντρίγκε τώρα, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ασχολούμαστε και μιλάμε για πολλαπλές κρίσεις. Πρέπει όμως να εντοπίσουμε τα κεντρικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν εάν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει σταθερή. Εάν θέλουμε να έχουμε μια Ένωση Ευρωπαίων. Νομίζω ότι τα δύο κεντρικά προβλήματα είναι η κρίση των ε, προσφύγων και η ε, καταπολέμηση της ανεργίας στην Ευρώπη. Πρέπει τα δύο αυτά προβλήματα να τα δούμε ε, ταυτόχρονα και μαζί να επιληθούν. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω τρεις πρωτοβουλίες, μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες να εκινηθούν, ώστε να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις απασχόλησης κυρίως για τους νέους σε τρεις, ε, με τρεις βασικούς στόχους προς επίτευξη. Να έχουμε πραγματικά ευρωπαϊκά σύνορα, να προσαρμοστούν οι κοινωνίες μας στην ένταξη των προσφύγων και να την επιδιώξουν ενεργά και να συνεργαστούμε με τις χώρες προέλευσης για να διαχειριστούμε τις ροές προσφύγων για να υπάρξουν σταθερά ευρωπαϊκά σύνορα, ξέρουμε ότι αυτό απαιτεί, είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, γιατί απαιτείται προσωπικό, λογισμικό, διοργάνωση λογιστικές υποδομέ. Χρειάζεται οι πολίτες μας να είναι σε επαγρύπνηση. Χρειάζεται σχεδιασμός θεσμικός και πολιτικός. Και έπειτα εάν υπάρξει κατάλληλη συνεργασία, πολλοί νέοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μια τέτοια ε, ενέργεια, σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Τέτοιου είδους προτάσεις πρέπει να, να υποβληθούν τώρα. Ευχαριστούμε η κυρία Αλβιόλ Κουσμάν. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σήμερα στην Ολομέλεια ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούγκερ, ο κύριος Αβραμόπουλο, Επίτροπο για τη μετανάστευση και ο κύριο Τάσκ, προεδρεύουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έπρεπε να παρετηθούν, να παρετηθούν για την αποτυχία τους να διαχειριστούν την προσφυγική κρίση, να παρετηθούν εξαιτίας της πρότασης για 160.000 μετανάστες και την μετακατάστασή τους που κατέληξε σε 162. Να παρετηθούν γιατί από τη δικιά τους την ευθύνα έχουν πνιγεί τόσοι άνθρωποι στη Μεσόγειο και τόσοι άλλοι ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στους καταβλισμούς. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ένας χώρος με έλλειψη αλληλεγγύης, ένας χώρος γεμάτο σκληρότητα. Τρία εκατομμύρια όμω υποσχέθηκε στην Τουρκία για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Τρία δι. για, την, ε, για τη θέση της Ευρώπης. Στα χέρια δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δίνει τρει φορέ παραπάνω χρήματα για την καταστολή στην Τουρκία από ό,τι για ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λούντκρεν τώρα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, είναι μια χρονιά γεμάτη αποτυχίες που πέρασε και τώρα έχουμε μια νέα χρονιά με πολλές δυνατότητες για νέες αποτυχίες. Έχουμε διαπιστώσει τι έχει γίνει με την μετανάστευση, πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα εξαιτία των αριθμών. Και βλέπουμε επίσης και νέες τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε διαστάσεις μάλιστα που ποτέ δεν είχαμε δει ξανά στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν τίθεται σε αμφισβήτηση από πολλούς. Στη χώρα μου πολλοί ρωτούν πρέπει να πληρώνουμε εμείς για να είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Τάσκ πληρώνονται. Αναρωτιέται ο κόσμος πόσα πληρώνονται για αυτή τη δουλειά. Πώς μπορεί κανείς να φανταστεί ότι εσείς εκπροσωπείτε τους Ευρωπαίους πολίτες. Κύριε Άτκινσον. Το Δεκέμβριο οι βιασμοί, σεξουαλικές παρενοχλήσεις και σεξουαλικές επιθέσεις φάρους των γυναικών ήταν στην ημερήσια διάταξη. Τώρα επανέρχονται λόγω της στάσης της Γερμανίας επέναντι στο θέμα αυτό. Έχουμε μαζικές ε, παρενοχλήσεις λόγω της ε, εισρωής, μαζικής εισρωής προσφύγων. Στο σχολείο τα κορίτσια πέφτουν θύματα παρενόχλησης στη Γερμανία και την Αυστρία. Οι Βαβαροί αποφασίζουν να στείλουν τους ε, ε, πρόσφυγές τους μέσα σε λεωφορεία στην κυρία Μέρκελ, η οποία τους στέλνει πάλι πίσω. Και αυτό άδικο για τους ετούντες στο άσυλο. Είχατε πει θα δεχθείτε 100.000. Τώρα σας φτάσανε κυρία Μέρκελ 1,2 εκατομμύρια. Τους δίνετε διαβατήρια. Αυτό σημαίνει με πολυπλησιαστικούς όρους έως και 10 εκατομμύρια επιπλέον άτομα που θα θελήσουν να φτάσουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο για να καταλάβουν περιοχές ε, με τον πληθυσμό που θα αναπτύξουν ισοδύναμες με αυτές ε, της δικής μου εκλογικής περιφέρειας, παραδείγματι. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν βοήθεια στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται τη Βόρεια Αφρική για να μπορέσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μια σύγκρουση πολιτισμών. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, ένα λεπτό και 30. Κύριε Πρόεδρε, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές συνεχίζουν αμύωτες και μάλιστα σε αναλογία δύο μετανάστες προς ένα πρόσφυγα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των αερογραμμών της Τουρκίας οι οποίες με 40 ευρώ μετακινούν χιλιάδες μετανάστες από τις χώρες του Μαγκρέπ και, το Μαρόκο με μοναδικό σκοπό να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι γνωστό ότι αυτές οι χώρες δεν χρειάζονται βίζα στη γειτονική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Οι παράνομοι διακινητές συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι. Μόνο στις τρεις τελευταίες εβδομάδες του 2016 77 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο, μεταξύ των οποίων και πάρα πολλοί νέοι και παιδιά. η πραγματική λύση είναι ο τερματισμός των συγκρούσεων στη συρία η επιστροφή των προσφύγων στις αιστείες τους η ασφαλής παραμονή στα σπίτια τους. λύση δεν μπορεί να είναι με τείχη μέσα στα εθνικά σύνορα των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης. χρειάζεται αλληλεγγύη και προστασία των εξωτερικών συνόρων της ευρωπαϊκής ένωσης των εξωτερικών συνόρων των λαών της ευρώπης. σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δύο λεπτά, Φλέκενστάιν. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είναι όλο και πιο εκρηκτική η κατάσταση και στη Γερμανία όλο και πιο εκρηκτική γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν είμαστε θέση να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και βέβαια δείχνουμε το δάχτυλο της Βρυξέλλες, όχι της πρωτεύουσας των κρατών μελών. Και εμείς έχουμε αυτή την ε, καταραμένη υποχρέωση να αποδείξουμε ότι δεν φταίμε εμείς. Είδα η Γερμανή οι Υπουργοί, ε, από το κόμμα του συνοδέλφου Ρέγνερ, Βέγνερ, σηκώνουν το ανάστημα στην κυρία Μέρκελ και λένε ότι θα πρέπει να κλείσουν τα σύνορα ή να ορίσουμε κάποια σχέδια. Με το κλείσιμο των συνόρων όμω δεν λύνονται τα προβλήματα, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται. Αντιθέτως, δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα. Για αν θέλουμε όμως να πείσουμε, θα πρέπει να προσφέρουμε περισσότερα στις χώρες μας από όσα προσφέρουμε φερειπίν με τον κύριο Τζοστκατ που λέει ότι κάναμε δεσμεύσεις, αναλάβαμε ε, δεσμεύσει, ε, είχαμε επικοδομητική συζήτηση με τον κύριο Κάμερον, ε, πρέπει να εντατικοποιηθεί η εσωτερική αγορά, να ενισχύσουμε την ενεργειακή αγορά κτλ. Ξέρουμε πολύ καλά όμως τι θα συμβεί από εκεί και πέρα και στο βαθμό αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Ούτε έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου χρειάζεται πια. Μα λέτε ότι ασχοληθήκατε πολύ καλά, σα πιστεύουμε. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τούσκ, ίσως θα ήταν καλή λύση να του κλείσετε όλου μαζί στο ίδιο δωμάτιο, Όπω γίνεται για την εκλογή του Πάπα. Σε ένα δωμάτιο το κονκλάβιο και να μην βγουν έξω αν δεν έχουν βρει λύση. Το να συνομιλούν ε, στο Συμβούλιο κάθε δύο μήνε ε, να βγάζουν συμπεράσματα για να πούν ότι τελικά δεν υπάρχει καμία λύση, δεν χρειάζεται πια για μα ακόμη φράση, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, για τον τρόπο με τον οποίο επιτελέσατε ένα πολύ δύσκολο έργο χτες. Χρειαζόμαστε δημοκρατία και όχι ε, Poland bashing. Δεν θέλουμε να καθιβρίζεται η Πολωνία, δεν χρειάζεται αυτό. Και το διαχειριστήκατε πολύ καλά. Κύριε Φλέκενστάιν, έχετε μπλε κάρτα. Σας ευχαριστώ που ξεπεράσετε τον χρόνο σας. Έχετε μπλε κάρτα, με ακούτε. Δεν, ξέρετε ποια είναι η ερώτησή μου, αλλά... Ο, λέτε το ναι. Ο συνάδελφος παρακαλώ να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Φλέγκενστάιν. Θέσατε ένα αμφιβόλο τις ε, δεσμεύσεις και τις επενδύσεις για την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα. Εάν δεν υπάρχουν έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα, τι έχετε να προτείνετε ως ε, εναλλακτική. Γιατί εύκολα επικρίνετε τους άλλους, αλλά δεν μας λέτε εσείς, σοσιαλιστές, τι θέλετε να κάνετε. Η απάντηση των σοσιαλδημοκρατών είναι η απάντηση που έχει δώσει το κοινοβούλιο μας. Πρέπει να προστατεύουμε και να ελέγχουμε τα εξωτερικά σύνορα. Ωστόσο, πέραν αυτού, πρέπει και εύλογα να σταματήσουμε να καταστρέφουμε το Σέγγεν. Αυτό είναι το καθήκον των Πρωθυπουργών, των ηγετών των κρατών που θα πρέπει να επιτελέσουν και πια να συνομιλήσουν μεταξύ τους για να βρουν λύσεις συγκεκριμένες για το τι πρέπει να συμβεί. Και να μπορεί ο κάθε Ευρωπαίος στο Σέγγεν μέσα να αισθάνεται σαν στο σπίτι του. Γιατί αν κλείσουν τα σύνορα του Σέγγεν, τότε και το Σίγεν δεν θα χρειάζεται, αλλά ούτε και η συζήτηση που κάνουμε. Κυρία Βουίλμοντ, ένα λεπτό και 30. Ενάμιση μου είπανε. Η καρδιά μου λέει ότι πάλι συζητάμε εδώ ένα πρόβλημα που δημιουργεί ο Ντέιβιτ Κάμερον αντί τις πραγματικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο σίγουρα οι ηγέτες ένιωσαν το ίδιο. Πρέπει όμως να γίνει αυτό, όχι γιατί στηρίζω τι διαπραγματεύσει του Κάμερον, δεν έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες αυτό και εγώ. Για παράδειγμα, πού είναι οι προτάσει όσον αφορά την νομοθεσία για τους εργαζόμενους, τους αποσπασμένους, για τις συνθήκες εργασίας τους. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ε, προτάσεις που ζημιώνουν και δεν βρίσκονται πια στο τραπέζι. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε γιατί αυτό βλέπουν σαν όφελος ή όχι οι Ευρωπαίοι. Συνεπώς, πώς θα συζητήσουμε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πρόκειται για τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζει τα εργασικά δικαιώματα η Ευρώπη. Και για ορισμένους είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Οι επιχειρήσεις έμεσα ή άμεσα εξαρτώνται από τις σχέσεις με την Ευρώπη. Οι εργαζόμενοι επίσης για όλους αυτούς με τίποτα δεν ε, πιστεύουν ότι θα ήταν καλύτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει συμφωνία και πρέπει να υπάρξει γρήγορα. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο Βρετανικό δημοψήφισμα και να πάψει αυτή η αβεβαιότητα και για την Μεγάλη Βρετανία και για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ναι, ένα μισή λεπτό είχατε πράγματι κυρία Βίλμοντ, λέει η Πρόεδρος, η κυρία Τόγια τώρα. Ένα λεπτό. Οι πολλαπλές κρίσεις που έχουν πλήξει την Ευρώπη οδηγούν σε αποσάρθρωση του συστήματο. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Όπω είπατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ, ό,τι περνάει από το χέρι σα για να σώσετε την Ευρώπη, να την κρατήσετε ενωμένη. Θέλουμε την Ευρώπη του σήμερα και του μέλλοντο. Γι' αυτό εμεί, οι Ιταλοί, ε, το Κοινοβούλιο και η κυβέρνησή μα πρέπει να δώσουμε τι κατάλληλε αποκρίσει. Πρέπει να κάνουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί για τη μετανάστευση. Πρέπει να προχωρήσουμε με την ευηλεξία και την ανάπτυξη και τι θέσει εργασία. Ε, πρέπει να είμαστε πιο αλληλέγγυοι και πιο προοδευτική στην Ευρώπη. Ω Ευρωπαϊστέ ε, και φίλοι είμαστε φιλόδοξοι. Ε, έχουμε ένα πρόγραμμα ανάκαμψη τη Ευρώπη. Δεν θέλουμε να αμφισβητείτε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, απλώ να είμαστε συνεπεί ω προ τι δεσμεύσει μα και τι υποσχέσει που έχουμε δώσει. Μεταξύ άλλων, να πούμε ε, ότι ο κύριο Βέμπερ. Δεν ξέρω ποιο είναι για να μα λέει τι συμβαίνει στην Ιταλία. Αλλά όταν μιλάει για μα και την κυβέρνησή μα, πάντοτε σφάλει. Είναι πολύ εύκολο ε, να κάνει τέτοια επικριτικά σχόλια. 30 δευτερόλεπτα. Ε, η Ευρώπη πιο πολύ κινδυνεύει εξαιτία του ιδίου και των φίλων του με τι ιδεολογικέ του ε, ε, ακαμψίε παρά ε, εμεί με τι ανισότητε των πολιτών που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, εργασία και κοινωνική ατζέντα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Γκαρσία Πέρες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Τούσκ όταν μίλησε είπε ότι η Ευρώπη είναι περισσότερο ισχυρή από ό,τι πιστεύουμε. Και εγώ θέλω να του πω ότι ακριβώς αυτό είναι και το πρόβλημα, η έλλειψη αξιοπιστίας. Γιατί ακόμα και εμείς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα και στηρίζουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο, μερικές φορέ δυσκολευόμαστε να το εξηγήσουμε και να το δικαιολογήσουμε. Σήμερα δεν είμαστε πρωτοσέλιδο. Παρόλα αυτά υπάρχει μια πραγματικότητα που πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε. Οι εθνικές κυβερνήσεις τι κάνουν για να πάρουν τις χιλιάδες τους πρόσφυγες οι οποίοι σε ακραίες θερμοκρασίες ζουν σε καταβλισμούς. Μπείτε στη θέση τους. Μπορείτε να σκεφτείτε να ήταν τα παιδιά μας σε αυτή την κατάσταση τάπα στο Συμβούλιο, τάπα στις εθνικές κυβερνήσεις. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Οι χώρες πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα προβλήματα είναι πολλά και οι λύσεις επίγουν και είναι αναγκαίο να βρεθούν. Ευχαριστούμε κυρία Ιώτοβα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιούνκερ για τις προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρει μια λύση στο προσφυγικό. Όμως θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αναφερθήκατε στο μέλλον. Το Συμβούλιο όμως, αυτό ακριβώς δείχνει το ότι μιλάμε για το μέλλον, ότι έχει κάνει λίγα μέχρι τώρα. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να κλείσουν τα σύνορά μας. Θέλουμε να έχουμε ένα νέο οργανισμό που θα προστατεύει τα σύνορά μας και θα καλύπτει μόνο το Σέγγεν. Όμως όχι όλα τα εξωτερικά σύνορα, έτσι δεν είναι. Γιατί όμως. Το έχω ρωτήσει αλλά δεν έχω πάρει απάντηση. Όσον αφορά τη συνεργασία με την Τουρκία επίσης δεν έχουμε απάντηση. Από ό,τι φαίνεται λίγα έχουν επιτευχθεί και υπάρχουν και πάρα πολλοί άγνωστοι παράγοντες όσον αφορά την βοήθεια που θα προσφέρει η Τουρκία εθελοντικά. Το θέμα... Ευχαριστούμε κυρία Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι τελευταίες ημέρες έδειξαν ότι η διάσωση της Ευρώπης μπορεί να γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μία μέθοδο τελείως καινούρια. Τη διάσωση με ίδια μέσα. Αυτό θέλω και να σχολιάσω. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έλαβε δύο επίσημες δεσμεύσεις. Πρώτον, να δημιουργήσει μια κοινή πιστοτική γραμμή, κάτι που να προβλέπει, όπως προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, και σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει χρηματοδότηση από το κοινό Ταμείο Διάσωση. Εδώ, πριν αρχίσουν να ισχύουν όλα αυτά, έπρεπε να προβλεφτεί αυτό ο μηχανισμό και υπήρχε μια τέτοια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία είχαν συμφωνήσει πέντε πρόεδροι. Αλλά κι άλλη μια συμβαστική λύση δεν επετέχθη. Αυτή του 2012 και τη εποχή του κυρίου Ρομπόη. Όταν υπήρχε ένα ενιαίο μηχανισμό ε, διάσωση, ο οποίο θα εξασφάλιζε και την ε, ε, προάσπιση των στοιχείων των ενεργητικού των τραπεζών. Εδώ λοιπόν είδαμε για άλλη μια φορά να μην επιτυγχάνεται αυτή η συμφωνία. Ελπίζουμε το 2017 τουλάχιστον το Συμβούλιο να κάνει όσο έχει υποσχεθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έκλεισε έτσι ο κατάλογο των αγορητών. Περνάμε τώρα στην... των εγγεγραμμένων στη λίστα των αγορητών. Περνάμε τώρα στην διαδικασία Η κυρία Σπυράκη, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε Γιούγκερ, δύο είναι οι όροι κλειδιά για την αντιμετώπιση της πιο επίγουσα κρίσης από τις κρίσεις που βιώνουμε η κρίση του μεταναστευτικού χρειάζεται εφαρμογή των δεσμεύσεων των κρατών μελών και χρειάζεται και επίβλεψη των συμφωνιών για την εφαρμογή τους με τις τρίτες χώρες. σε ό,τι αφορά το πρώτο θα τολμούσα να πω ότι είναι η ώρα να σκεφτείτε πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα μηχανισμό κυρώσεων για τη μη εφαρμογή της υποχρεωτικής μετεγκατάστασης στα κράτη μέλη πιστεύω βαθιά ότι η ανισορροπία της συνεισφοράς στη μεταναστευτική κρίση είναι θριαλίδα στο θεμέλια της ένωσης. δεν μπορούν οι μικροί οι αδύναμοι αυτοί που μαστίζονται από την κρίση να σηκώνουν δυσανάλογα βάρη με τους ισχυρούς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τις τρίτες χώρες είναι ανάγκη η τουρκία να κάνει πολύ περισσότερα βήματα. μόνο τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες έφτασαν στην ελλάδα από την τουρκία 30.000 άνθρωποι εκ των οποίων οι ελάχιστοι ήταν πρόσφυγες. κυρίως δεν επαναπροωθούνται και οι παράτυποι μετανάστες. χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό έχει λήξει ο χρόνος σας ο κύριος Κύριος Τίμπορ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητήσαμε και ακούσαμε προσεκτικά όσα μας είπε το Συμβούλιο και η Επιτροπή και πραγματικά αρχίζω να αναρωτιέμαι τι κάνουν εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολομέλεια και πρέπει να απολογηθούμε για σφάλματα που έχουν διαπράξει στα κράτη-μέλη, σε άλλο θεσμικό όργανο. Δηλαδή, επικροτήσαμε την δήλωση υποδοχής προσφύγων από την καγκελάριο Μέρκελ. Όμως, μια καγκελάριος ή ένας καγκελάριος της Γερμανίας έχει δικαίωμα και έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Διότι βλέπουμε στη συνέχεια κάποια κράτη να σηκώνουν και να υψώνουν ε, σύνορα και φραγμούς και κάποιοι άλλοι όχι. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την οδό των Βαλκανίων. Εκεί πρέπει να πούμε όχι και όχι στις μεμονωμένες πολιτικές κινήσεις των κρατών Πρέπει να δράσουμε από κοινού. Ευχαριστώ εδώ για να αναλάβουμε και πάλι τον έλεγχο των πραγμάτων θα πρέπει να καθορίσουμε την μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης πως τώρα ήταν χειριστή. Όλοι οι πολιτικοί ηγέτες έλαβαν αποφάσεις δημιουργώντας προβλήματα που μας απασχόλησαν ακόμη για μήνες και θα μείνουν στην πλάτη μας για δεκαετίες. Θα πρέπει να επιστρέψουμε τι αρχέ του προβλήματο. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιε μεταναστευτικέ κρίσει χωρί να εφαρμόσουμε σωστά του νόμου. Ή θα έχουμε κατακλυσμό, θα πλημμυρίσουμε από ε, πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε την πολιτική του ασύλου για να προστατεύσουμε τα άτομα που κινδυνεύουν στι χώρε προέλευσή του, όμω δεν μπορούμε να σώσουμε ολόκληρο έθνο, Εάν συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε τόσους μετανάστες όπω του τελευταίου μήνε, θα ε, αλλάξουμε την ισορροπία τη Ευρώπη, την ασφάλειά μα για λόγους κοινωνική προστασία, λοιπόν. Πρέπει να εφαρμόζουμε σωστά του κανόνε, διότι μόνον έτσι θα μπορούμε να ε, επιτρέψουμε την ένταξη αντί να καταστρέψουμε την αρχή τη Ευρωπαϊκή ε, αλληλεγγύης. Το μεταναστευτικό είναι ένα ακόμη σοβαρό θέμα το οποίο δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε με εσφαλμένο τρόπο. Το άφησε να δημιουργηθεί, να διωγγωθεί και τώρα δεν έχει το θάρρο να το επιλύσει με τον προβλεπόμενο τρόπο. Η λύση του προβλήματο δεν είναι να υψώνουμε στα σύνορα τείχη ούτω ώστε να καταργούμε στην πράξη τη συνθήκη Σέγγεν. Η λύση του προβλήματο είναι να σταματήσουν οι πόλεμοι που δημιουργούν πρόσφυγες και μετανάστες. μέχρι τότε όμως η λύση αυτή βρίσκεται στην τουρκία. εκεί πρέπει να εγκατασταθούν τα κέντρα διαλογής ε, προσφύγων τα hot spots ούτως ώστε να μην τους επιτρέπουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες να έρχονται στην ελλάδα. επίσης εάν υπάρχει μια χώρα στην οποία πρέπει να εγκατασταθεί η ευρωπαϊκή δύναμη αυτή είναι η τουρκία ούτως ώστε η δύναμη αυτή να μην επιτρέπει στο μεν επίσημο κράτος να εκμεταλλεύεται τους παράνομους μετανάστες για να επιδιώκει να επιλύει εθνικά του θέματα ούτε και στους διεφθαρμένους κρατικούς φορείς να κερδοσκοπούν εις βάρος αυτών των δυστύχων ανθρώπων. Απ' την άλλη πλευρά οι ελληνικές δυνάμεις ακτοφυλακής μπορούν και να επιβλέψουν και να επιτηρούν τα σύνορα της Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Εκτιμάω απόλυτα την πρωτοβουλία όσον αφορά την κοινή φύλαξη των συνόρων. Απόφαση που λήφθη το Δεκέμβριο. Από την άλλη μεριά όμως απογοητεύομαι, γιατί η συμφωνία αυτή αναβάλλεται μέχρι τον Ιούνιο του 2016 από ό,τι φαίνεται. Στη συζήτηση ακούσαμε ότι οι περισσότεροι ευρωβουλευτές θέλουν να εγκριθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η πρωτοβουλία. Κάνω έκκληση λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς είσαστε αρμόδιοι, υπεύθυνοι και καταλαβαίνετε ότι θα σας στήριζε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν το κάνατε. Γι' αυτό η συμφωνία πρέπει να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τι εμποδίζει στο επόμενο συμβούλιο, ακόμα και ένα έκτακτο συμβούλιο που θα μπορούσε να οργανωθεί για το Φεβρουάριο, να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία ώστε να αρχίσει η κοινή αυτή προστασία των συνόρων. Ευχαριστούμε τέλησε, τέλειωσε το Καρσδιάι. Εσείς τώρα, Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, καταλαβαίνω αυτούς που δηλώνουν κουρασμένοι από τις επαναλήψεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Το καταλαβαίνω και ακούσαμε από τον κύριο Τάσκ ότι οι χώρες μέλη δεν έκαναν πράξη τις αποφάσεις που πήραμε. Οι χώρες φταίνε, όχι όλες, αλλά ένας μεγάλος, εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός, θα έλεγα. Γι' αυτό και κάθε τόσο επαναλαμβάνουμε τις ίδιες εκκλήσεις. Δεύτερον, κατάλαβα από κάποιες παρεμβάσεις σας ότι πιστεύετε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοτείται παρκώς. Και ακολουθώντας, μάλλον είπατε πολύ από εσάς ότι η, Ευρώπη, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει αυτά που πρέπει. Εγώ όμως από ό,τι βλέπω, μάλλον το αντίθετο θα έλεγα, ότι εμείς όντως κάνουμε αυτά που χρειάζεται για να προσανατολιστούμε προς την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Το 2014 ήδη ξεκινήσαμε με το επενδυτικό πρόγραμμα με τα 315 δισεκατομμύρια. Δεν σας έχει ξεφύγει αυτό, το ξέρετε. Και ήδη 40 δις έχουν ήδη κινητοποιηθεί με 47 μεγάλα προγράμματα υποδομών, 11 στην Ιταλία και 7.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ασχολείται με το θέμα της ασφάλειας, με το θέμα της ενέργειας. Όλες οι δράσεις που έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά, ψηφιακή αγορά κτλ. Οπότε δεν βλέπω γιατί αμφισβητείτε την πορεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λέτε ότι δεν έκανε τη δουλειά τη τον πρώτο χρόνο αφότου ανέλευε τα καθήκοντά της. Τώρα τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν στην συζήτηση σήμερα Κάποιος φιλικά μου είπε ότι θα έπρεπε να παρετηθώ επειδή δεν μπορέσαμε να λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προσφυγικό. Μα δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε. Οι δράσεις οι οποίες αποφασίστηκαν τώρα πρέπει να τεθούν και σε εφαρμογή, να υλοποιηθούν. Κατά τα άλλα, Πρόεδρε, δεν έχω παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βινκέρ και τώρα για να ολοκληρώσουμε ο πρόεδρος, κύριος τους πρόεδρος του Βουλίου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καταρχάς έχετε απόλυτο δίκαιο. Έχουμε πρόβλημα στην υλοποίηση αυτή τη στιγμή. Και σε σχέση με την κρίση τη μεταναστευτική, αναμφίβολο, ζούμε κρίσιμη περίοδο. Και αυτό όχι μόνο όσον αφορά την υλοποίηση των αποφάσεών μας, αλλά και γιατί είναι ίσως η πρώτη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για κρίσιμη στιγμή για το πολιτικό σύστημα το ίδιο στην Ευρώπη. Η Ευρώπη στηρίζεται ε, στο αξίωμα ότι όλοι μας, όλα τα κράτη-μέλη, είμαστε διατεθειμένοι να δράσουμε με καλές προθέσεις και να σεβαστούμε, να σεβαστούν τις κοινέ αποφάσεις. Πάνω σε αυτό στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αυτό δεν έχει λόγο ύπαρξης αυτή η συνεργασία. Σε αυτό έχει έχετε απόλυτο δίκαιο. Η κρίσιμη στιγμή σήμερα λοιπόν είναι ότι δεν έχω δυσκολία στην πραγματικότητα να επιτύχω συμβιβασμούς στο δικό μας το επίπεδο, στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Των αντίον. Παρά είναι εύκολο, εύκολη η επίτευξη των συμβασμών. Γιατί? Γιατί την επόμενη μέρα δεν είναι κανείς διτεθειμένος να σεβαστεί τις κοινέ αποφάσεις. Και αυτή είναι η κρίσιμη. Αυτό δείχνει την κρισιμότητα μάλλον ε, της κατάστασης, όχι μόνο για τη μετανάστευση, αλλά και για την Ευρώπη την ίδια ως πολιτικό οργανισμό. Είναι πολύ δύσκολο να καλέσουμε σε πειθαρχία τα κράτη-μέλη. Και θα πω το εξής και συγχωρέστε μου την ε, αμεσότητα. Αν αυτή η βασική αρχή, ο πρώτος κανόνας δηλαδή πρωταρχικός, ότι οφείλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και τους κανόνες, τις αποφάσεις που λαμβάνουμε, αν αυτή η βασική αρχή δεν τηρείται, στο πρώτο από το πρώτο ήδη στάδιο έχουμε τεράστια προβλήματα ως προς την υλοποίηση της δουλειά μας. Γι' αυτό και δεν έχω να πω ούτε ευχαριστώ ούτε τίποτα άλλο στην Επιτροπή, ζητώντα συγγνώμη για την ε, ε, αγένεια. Είναι αυτή η σκληρή αλήθεια. Η Ευρώπη ως οργανισμός και τα κράτη-μέλη δεν ήταν έτοιμοι, δεν ήταν έτοιμα να αντιμετωπίσουν αυτή την τελείως νέα σε κλίμακα, σε νούμερα κρίση τη σχετική με τη μετανάστευση. Σωστό είναι αυτό. Με τη δική σας την εκτίμηση όσον αφορά τη συζήτηση για τα εξωτερικά σύνορα δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω και στο συγγνώμη, αλλά όταν συζητούμε τα εξωτερικά σύνορα, την ενδύση δηλαδή των εξωτερικών σύνορων, πρόκειται για μια καινοτόμο, ε, καινοφανή μάλλον ιδέα. Θα θυμάστε ίσως, γιατί εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, ότι στην αρχή της συζητήσεως για τη μεταναστευτική κρίση, αλλού δινόταν ο τόνος. Άλλο θέμα ήταν ε, τη επικαιρότητα και όχι τα εξωτερικά σύνορα. Σε αυτό αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για τα όσα κατάφερε η Επιτροπή στο θέμα τη ενίσχυση των εξωτερικών σύνορων και την ε, καινοφανή αυτή ιδέα για μια κοινή συνοριοφυλακή για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων στην Ευρώπη. Κάποια από τα στοιχεία αυτής της ιδέας παραμένουν ακόμα αμφιλεγόμενα για ορισμένα κράτη-μέλη για διαφορετικούς λόγους. Πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση. Θα πρέπει δηλαδή να τα πείσουμε, να τους εξηγήσουμε και να πείσουμε ότι μπορεί να είναι νέα, μπορεί να είναι αμφιλεγόμενη, αλλά απόλυτος απαραίτητη αυτή η λύση. Αυτό που χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα είναι νομίζω να προχωρήσουμε στην επίλυση κάποιων προβλημάτων το ταχύτερο δυνατό. Εξού και η συνεδρία του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου θα είναι αφιερωμένη στο Βρετανικό, ελπίζοντας ότι θα είναι και η τελευταία η σχετική με το ζήτημα της Βρετανίας. Και βέβαια ταυτόχρονα θα αξιολογήσει, θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της υλοποίησης των μέτρων των σχετικών με την μετανάστευση και τα σχετικά με την Τουρκία και το πρόγραμμα δράσης για την Τουρκία. Το επόμενο Συμβούλιο του Μαρτίου θα είναι αφιερωμένο και αυτό, αλλά όχι μόνο, όχι αποκλειστικά, στη μεταναστευτική κρίση. Ε, διατυπώθηκαν κάποιες ερωτήσεις σχετικές με την Πολωνία. Όπως είπα νωρίτερα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μερικέ ημέρε, σε μια συνάντηση με τις πολιτικές ομάδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαίωμα και υποχρέωση να προβεί σε σκληρό, σε ειλικρινή και ε, απερίφραστο διάλογο σε σχέση με τις ε, ενδεχόμενες παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων. Μην περιμένετε όμως να είμαι και περιχαρής όταν ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία για την Πολωνία. Είμαστε απόλυτος βέβαια. Όχι, παρακαλώ να το κατανοήσετε. Ότι βρίσκομαι σε δύσκολη θέση. Είναι δύσκολο για μένα αυτό και ξέρω ότι δρά καλόπιστα η Επιτροπή, δεν έχω καμιά αμφιβολία περί αυτού. Βεβαίως και μπορούμε να συζητούμε κάποια μέτρα μεθόδους, αποφάσεις της Επιτροπής που θα μπορούσαν να ήταν οι πιο σκληρές, οι πιο ήπιες, μπορεί να συζητούνται και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και θέματα σε σχέση με τη στάση και τις δηλώσεις επιτρόπων ή διαδικαστικά θέματα που θα μπορούσαν διαφορετικά να ε, διαμορφώθουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελήφθη μια απόφαση. Η Επιτροπή έλαβε την απόφαση αυτή. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η απόφαση αυτή είναι η βέλτιστη και την αποδέχομαι και την υποστηρίζω απολύτως. Μην αναζητείτε συγκρούσεις ή ρήγματα στη σχέση μεταξύ των θεσμών. Ειδικά για το θέμα αυτό. Είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και σε σχέση με αυτό. Και όταν έρθει η ώρα για την ε, συζήτηση για την Πολωνία, πολύ σύντομα ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προεδρεύον του Συμβουλίου. Διακόπτω για μερικά λεπτά.